το βράδυ αρχίζει η προθεσμία για τι διαπραγματεύσει. Τελευταία ανακοίνωση και μετά θα δώσω το λόγο στου συναδέλφου που το ζητούν. Θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου, ο πρόεδρο Ταγιάννη, αύριο θα εγκρίνει δύο πράξει σύμφωνα με τη συνήθη ε, νομοθετική διαδικασία και το άρθρο 78 του κανονισμού ο τίτλος των πράξεων αυτών θα δημοσιευθεί στα πρακτικά. Σας ευχαριστώ για την ε, υπομονή σας. Πριν έρθουμε στη διάταξη των εργασιών, τρεις συνάδελφοι ζητούν το λόγο. Ο κύριος Φρουντσούλικα για διαδικαστικό. Τρεις είναι συνάδελφοι. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, στις 20 Νοεμβρίου στο Κίεβο έλαβε χώρα ένα φόρουμ εθνικών μειονοτήτων στην Ουκρανία συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της ρουμανικής, βουλγαρικής, ε, σλοβακικής μειονότητας μεταξύ άλλων Τατάρων και Εβραίων για τη συζήτηση για το νέο νόμο που απαγορεύει στις εθνικές μειονότητες να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους ε, στη γλώσσα τους σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, σε όλες τις βαθμίδες. Άρθρο 7. Και ε, το πολιτικό κίνημα Σφοποντά στην Ουκρανία ε, διέκοψε αυτή τη διαδήλωση. Παρακαλώ να λάβει θέση το Κοινοβούλιο για αυτά τα σημαντικά ζητήματα. και γιατί οι Ουκρανικές αρχές ανέχονται τέτοια πράγματα. Είναι συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουκρανία και θα πρέπει να σέβεται και να συμμορφούνται με τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές και να τις προωθεί. Μεταξύ αυτών είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα των ε, εθνικών μειονοτήτων στη χώρα που έχουν δικαίωμα, όπως γνωρίζετε, στην εκπαίδευση στη μητρική τους γλώσσα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Σημειώνουμε τα σχόλιά σας. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Σουίτσα. Παρακαλώ, διαδικαστικό. Uh, I would like to speak in my mother tongue. Θα ήθελα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να ενημερώσω το Κοινοβούλιο ότι το Κροατικό Κοινοβούλιο διέκοψε την ε, συνεδριασή του, όπως και το Κοινοβούλιο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν έξι Κροάτες ε, της ε, Βοσνίας στο δικαστήριο της Χάγης, οι οποίοι καταδικάστηκαν. Ένας εξ αυτών υπήρχε μια δόση δηλητήριο όταν ανακοινώθηκε η απόφαση του δικαστηρίου και πέθανε. Θεωρώ πως ε, εφόσον ε, τα κοινοβούλια αυτά διέκοψαν ε, την συνεδρίασή τους θα έπρεπε τουλάχιστον να σας ενημερώσω για το τι συνέβη πέρα από τα γεγονότα του πολέμου και διάφορα πράγματα που ακούγονται δεν ισχύουν. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ινετφέλτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όλοι ε, γνωρίζουμε πως οι πολιτικές ε, συζητήσεις ε, καμιά φορά γίνονται έντονες αλλά σοκαρίστηκα παρά το ότι αρκετά χρόνια στην πολιτική που είδα τις εικόνες ενός απαγχωνισμού διαδικτυακού έξι Πολωνών συναδέλφων. Χαίρομαι που αντέδρασε άμεσα ο κύριος Σταγιάννη και ζήτησε από την κυβέρνηση Πολωνίας να διασφαλίσει την ασφάλεια των έξι συναδέλφων και πράγματι ο Πρωθυπουργός Πολωνίας τα καταδίκιασε αυτά, είπε η Πρωθυπουργό. Αλλά ταυτόχρονα είπε, κοιτάξτε τη συμπεριφορά των Ευρωβουλευτών και πώς ε, δυσφημίζουν την Πολωνία και μάλιστα και ένα κομματικό τη φίλο για αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου έχει κάνει παρόμοια σχόλια για διάφορου βουλευτέ και για εμένα. Υπάρχει ελευθερία λόγου, αλλά ελπίζω να έχουμε λίγο σεβασμό και ο πρόεδρο κ. Σταγιάννη να πιέσει την πολωνική κυβέρνηση να μην διασφαλίσει μόνο την σωματική ακαιρεότητα των συναδέλφων αλλά να διασφαλίσει και την ελευθερία λόγου ακόμα και για πράγματα που δεν αρέσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ σημαντική αυτή δήλωση. Όπως ξέρετε ο κύριος Ταγιάννη έχει αναλάβει δράση και η λέξη σεβασμός νομίζω ε, είναι μια λέξη που πρέπει να ακούγεται συχνότερα. Ναι, σας... Κύριε Ντάτμουθ, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επί της ε, διαδικασίας ε, να ρωτήσω την κυρία Ίνετφελντ εάν ε, αυτά τα οποία λέει για την ελευθερία του λόγου ισχύουν και εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι μόνο εκτός. Αν μου επιτρέπετε θα απαντήσω εγώ και η απάντηση είναι ναι. Θα συνεχίσω τώρα το τελικό σχέδιο. Ορίστε. Κυρία Χάρμς, με συγχωρείτε. Όχι. Ναι, κυρία Χάρμς, ναι, δεν σας είδα. Θα επανέλθουμε στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να προσθέσω στα όσα είπε η συνάδελφος από την Άλντε ότι για εμένα ήταν πολύ ανησυχητικό αυτό το οποίο είδα στα κοινωνικά μέσα τις εικόνες δηλαδή πολλών συναδέλφων από την Πολωνία που δείχνουν τους ε, συναδέλφους απαγχωνισμένους. Δεν είναι κάτι το οποίο καλύπτεται νομίζω από την ελευθερία έκφρασης. Ε, πρόκειται για μια εγκληματική πράξη. Και αυτό το οποίο περιμένουμε από τους συναδέλφους ε, του προέδριου περιλαμβανομένου του αντιπροέδρου μας από την Πολωνία είναι όχι μόνο να απολογηθούν ε, λεκτικά αλλά να κάνουν κάτι για αυτή την υπόθεση η οποία είναι τρομερή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Χάρμς. Είναι σοβαρό πολύ το θέμα. Το έχουμε σημειώσει. Έχει εκφραστεί και η Ολομέλεια. Λοιπόν, ζητάνε και άλλοι συνάδελφοι τον λόγο. Τώρα δεν θέλω να γίνει συζήτηση για το θέμα. Θα δώσω τον λόγο όμως στον κύριο Καζουντεύσκη. Συνάδελφοι, οι πολωνικές αρχές ασχολούνται με το θέμα. Οι συνάδελφοι να μην ανησυχούν. Σας ευχαριστώ για αυτή την πληροφορία. Ο κύριος Βάγγελ, εμείς εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους διάφορους ε, συναδέλφους. Θα ήθελα να ζητήσω από το Κοινοβούλιο να δείξει αλληλεγγύη σε δύο πρώην μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρίσκονται στη φυλακή στην Ισπανία. Νομίζω ότι πρέπει να ε, εγκαταλείψουμε αυτή τη μας ε, την σιωπηρή συνωμοσία και να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει εκεί. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, ανέφερα το τελικό σχέδιο τη ημερήσια διάταξη υιοθετήθηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων στι 15 Νοεμβρίου με, σύμφωνα με το 149, το άρθρο 149 και τώρα θα αρχίσουμε διαβουλεύσει με τι ομάδε για να υποβάλουμε τι εξή ε, αλλαγέ. Δήλωση τη Επιτροπή για σήμερα για την απόφαση για τη δίκαιη φορολογία, το δεύτερο πακέτο αυτό αναβάλλεται. Δήλωση των θανατηφόρων πλημμυρίων στην Αττική, καθώς και η σχετική βοήθεια προστίθεται για αύριο κινητοποίηση του ε, περιθωρίου για το 2017 προστίθεται και η ψηφοφορία για την έκθεση κυρία Σαγκοράφα για την ε, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιβάνου αναβάλλεται. Υπάρχουν αντιρρήσεις, όχι, οπότε γκρίνονται και μια προσθήκη για αύριο. Η, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων υιοθέτησε την έκθεση ε, ασυλίας της κυρίας Φεράρα σύμφωνα με, τον, με το άρθρο 9.9 η έκθεση αυτή θα ψηφιστεί την Πέμπτη και η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με αυτέ τι αλλαγέ. Και έτσι τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο πρώτο σημείο τη ημερήσια μα διάταξη, που είναι η δημοσιονομική διαδικασία για το 2018 και έχουμε πρώτα στη σειρά τον πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, τον κύριο Αρτουή. Ε, ε,